Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nur noch. Ich darf. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας καλωσορίσω ξανά στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Έχουμε περάσει τώρα στην απαλλαγή άλλα όργανα. Γενικός εισηγητής είναι ο Τόμας Τεχόφσκι και έχετε αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία. Και μια πολύ καλή συνεργασία και καλές σχέσεις ε, σε ό,τι αφορά τις εργασίες της Επιτροπής μας. Εύχομαι λοιπόν το 2020 να συνεργαστούμε καλά έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε την απάτη και τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ άλλων. Είμαι υπεύθυνο λοιπόν εισηγητής για την απαλλαγή στα άλλα όργανα για το 2018. Είναι μεγάλη μου χαρά λοιπόν που βλέπω ότι το ελεκτικό συνέδριο αποφάνθηκε ότι τα άλλα όργανα λειτουργούν εύρυθμα και ότι δεν υπάρχουν σοβαρά συστημικά προβλήματα. Η ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για το 2018 λοιπόν αναφέρεται στα επιμέρους όργανα, σε εσωτερικούς ισολογισμούς και Βασισμένος στην έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου κατάρτισα την δική μου έκθεση. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης της έκθεσης ήρθα και εγώ ίδιο σε επαφή με εκπροσώπους από τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλω να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος και ικανοποιημένος σχετικά με τη χρηστή οικονομική διαχείριση στα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρηστή διοίκηση, υπήρξε βελτίωση διαφάνειας και δεν παρατηρήθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην, ε, στα οικονομικά. έγινε μια μεγάλη προσπάθεια εξυγχρονισμού και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ζητήσαμε για την έκθεση αρκετές πληροφορίες, λάβαμε πολλά στοιχεία, ε, Έχετε στη διάθεσή σας όλα τα σχετικά στοιχεία στα παραρτήματα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω ε, λέγοντας προς το Συμβούλιο ότι πρέπει να βρούμε μια συμβιβαστική λύση για τη ε, διαδικασία απαλλαγή. Συμβούλιο και Κοινοβούλιο πρέπει να καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό. Έχω συναντηθεί άτυπα με διάφορους εκπροσώπους του Συμβουλίου. Είχαμε μια καλή ε, συνεργασία, μια καλή επαφή και εύχομαι η πρόεδρος της Επιτροπής μας, κυρία Χολμάιρη, να βρει μια καλή λύση. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι θα καταφέρουμε να συνεννοηθούμε με το Συμβούλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, να πω ότι γνωρίζω πολύ καλά πως ε, υπάρχει μία νέα οργάνωση εντός του ελεκτικού συνεδρίου. Θα οδηγήσει αυτό, ελπίζω, σε καλύτερη διαχείριση του φόρτου εργασίας. Και ελπίζω να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ηλεκτρικού συνεδρίου και επιμέρους οργάνων. Στο ηλεκτρικό συνέδριο είδαμε αρκετές βελτιώσεις. Για παράδειγμα, έγινε προσπάθεια βελτίωσης των οργάνων εσωτερικού ελέγχου, τόσο για τις εκ των προτέρων όσο και για τις εκ των υστέρων ε, για τους ελέγχους. Σε αυτό βοήθησαν και οι αντίστοιχε οδηγίε. Όλαφ επίσης έδειξε πως κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για τη διεξαγωγή ελέγχων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εδώ να πω ότι καλωσορίζω τι προσπάθειες της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών για βελτίωση τη επικοινωνία Είναι, ήταν πιο συνεργατική, ήταν διαθέσιμη σε επικοινωνία και ένωσαν τις ε, διοικητικές τους υπηρεσίες για να πλουστευτεί το έργο τους και το δικό μας. Και είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία τους ε, θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Όλαφ, να πω ότι πρόσφατα καταρτίστηκε μία μυστική έκθεση σχετικά με το φόρτο εργασίας των υπαλλήλων. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή δεν σημείωσε καλές επιδόσεις στον τομέα αυτό και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για την χορήγηση της απαλλαγής να λάβουμε υπόψη το γεγονός αυτό. Ε, Όλαφ δεν ε, έχει θέσει τη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω να λάβουμε και εμείς αυτήν την έκθεση του Όλαφ. διότι φυσικά δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις συστάσει του όλα χωρίς να έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας. Ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητή πρέπει και εκείνος ε, να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Και σίγουρα τόσο όλα όσο και ο θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θα πρέπει να αναλάβουν ακόμα περισσότερε αρμοδιότητε, μεγαλύτερο φόρτο εργασία, χωρί την κατάλληλη χρηματοδότηση. Πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη στις, ε, στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και το γεγονός αυτό, ο μεγαλύτερο φόρτο εργασία. Διότι για να αυξηθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη υποδομή. Επίσης, έχει σημειωθεί πρόοδος και ως προς τις επιδόσεις σε θέματα προϋπολογισμού. Εδώ σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε πολλούς ε, τομείς. Όμως έχουν γίνει και διοργανικές ε, συμφωνίες για ενισχυμένη συνεργασία. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική μεταξύ όλων των οργάνων. Και η ανταλλαγή των πρακτικών θα πρέπει να γίνει συνήθεια. Αυτά λοιπόν από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προσθέσω κι εγώ με τη σειρά μου ότι χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα αποτελέσματα των ε, διαβουλεύσεων με το Συμβούλιο. Μαζί με τους ε, συντονιστές θα στείλουμε μια επίσημη επιστολή στη διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών για να λάβουμε διαπραγματευτική εντολή. Θα δούμε τι θα γίνει και αν το Συμβούλιο θα είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί. Ας προσπαθήσουμε έστω να δούμε τι θα γίνει. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη θα λάβει το λόγο η Ιζαμπέλ Γκαρθία Μουνιός ως κοιόδηση συγγήτρια για τα άλλα όργανα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πληρέστατη εργασία που έκανε για την εκπόνηση οκτώ εκθέσεων για αυτά, θεσμικά αυτά όργανα και σημειώνω και εγώ την ανησυχία που είχα και εγώ εκφράσει για το ότι στις τελευταίες οικονομικές χρήσεις μειωνόντουσαν οι ε, έρευνες ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Επομένως, το εύρος ε, και οι συστάσεις στην κατηγορία αυτή είναι περιορισμένες και δεν μας βοηθούν και τόσο πολύ. Μιλάω για τις έρευνες που κάνει το ελεγκτικό συνέδριο. Οι εκθέσεις, ωστόσο, οι ειδικέ εκθέσεις, ε, αντίθετα αυξάνονται. Και νομίζω ότι το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να κατανείμει με πιο σωμερή τρόπο τις προτεραιότητες. Τώρα, από εδώ και πέρα, παρατηρώ ότι εσείς, κύριε Σδεχόφσκι, έχετε προσθέσει αρκετές παραγράφους για να αναφερθείτε στην κατάσταση αυτή. Εγώ συμφωνώ απολύτως με το περιεχόμενο, ωστόσο είναι κάπως ε, διάσπαρτα και αυθαίρετα τα σχόλια. Παράδειγμα, ε, κάνετε αναφορά ε, στις εκθέσεις για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης σε δύο περιπτώσεις και για την ΕΟΚΕ ε, για, το, για τη διαμεσολαβήτρια ε, και το Συμβούλιο, αλλά όχι ε, παντού. Και κανονικά πρέπει να μπει στο κομμάτι που μιλάμε για το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ελεγκτικού συνεδρίου και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα δεν φταίνε καθόλου. Δεν ευθύνονται για αυτή την κατάσταση. Θα σας πρότεινα λοιπόν για τις παραγράφους αυτές να τις βάλετε στην έκθεση για το ελεγκτικό συνέδριο και να τις αφαιρέσετε από τα άλλα ή αλλιώς να μπουν παντού. Αν και νομίζω η πρώτη επιλογή είναι καλύτερη. Αν συμφωνείτε βέβαια. Μπορώ να καταθέσω και σχετικές τροπολογίες ή μπορείτε να το κάνετε απευθείας εσείς. Μπορούμε να το δούμε διμερώς. και ε, σε σχέση και με τις εξωτερικές, εξαιρετικές ε, σχέσεις συνεργασίας που λέτε, ορίστε που προσφέρομαι να γίνει πράξη αυτό. Κάτι άλλο που σκέφτομαι είναι μήπως θα ήταν μια καλή λύση το ελεγκτικό συνέδριο να διενεργήσει μια ειδική έκθεση για τα θεσμικά όργανα όπως κάνει για τους εκτελεστικούς οργανισμούς ή για τα ευρωπαϊκά σχολεία. Και ακριβώς στην διαγραμμή πλεύσης Νομίζω ότι καλό θα ήταν να γίνει και μια οριζόντια έκθεση για τα λοιπά θεσμικά όργανα ή γενικά για τους θεσμούς. Α, δεν μου είχατε βάλει χρονόμετρο, πρόεδρε. Α, να μιλάω πιο αργά. Α, ναι, απλά, εντάξει, αν δεν έχω χρονόμετρο, να μιλάω πιο αργά. Όπω κάναμε για του εκτελεστικού οργανισμού λοιπόν, ζωντανή έκθεση γίνει και για, τους, για τα θεσμικά όργανα. Γιατί έτσι ε, θα κάνουμε πιο έτσι, απλές τις ειδικέ εκθέσει, αφαιρώντα αυτά τα γενικά στοιχεία και ταυτόχρονα θα μπορούμε σε μία έκθεση και μόνη να πραγματευτούμε όλα αυτά τα οριζόντιου χαρακτήρα, ζητήματα τα οποία ενδιαφέρουν όλα τα θεσμικά όργανα, δηλαδή ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αναφέρθηκε ο συγητής, διοργανική συνεργασία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε για το ε, τρέχον οικονομικό έτος, αλλά ε, θα ήθελα να το προτείνω στην Επιτροπή μας, ε, το προτείνω στην Πρόεδρο, στους συντονιστές και στη Γραμματεία εν ώψη της προσεχούς οικονομικής χρήσης. Και κάποιες τροπολογίες, τις οποίες θα καταθέσω, ακόμα δεν τις έχω ολοκληρώσει, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να σημειώσουμε ήδη κάποια θέματα που με ανησυχούν όπως οι συμφωνίες ε, της ε, ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών με το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Το έχω ξαναπεί κατά το παρελθόν. Δεν νομίζω ότι είναι ισορροπημένε ε, αυτέ οι συμφωνίε σε βάρο των δύο επιτροπών των συμβουλευτικών. Σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο, χάνουν οι επιτροπέ 60 μεταφραστέ, οι οποίοι πηγαίνουν στη νέα διεύθυνση, στην υπηρεσία έρευνα, στο EPRS στο Κοινοβουλίο. Αυτές τις υπηρεσίες έρευνας μπορούν να τις αξιοποιήσουν οι δύο ε, συμβουλευτικές επιτροπές, αλλά πρέπει να καταργήσουν τη δική τους μεταφραστική υπηρεσία. Αυτό ήταν το τίμημα. Και επίσης πρέπει μετά να πάνε σε ε, πρόσληψη προσωρινών ε, υπαλλήλων, συμβασιούχων ή να κάνουν εξωτερική ανάθεση. Και μιλάμε για ε, τουλάχιστον ε, ένα εκατομμύριο ευρώ έξοδα επιπλέον για την εξωτερική ανάθεση σε μεταφραστές εξωτερικούς. Ε, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να, να δοθούν αλλού, εάν δεν είναι πολύ υψηλό ο λογαριασμός <clears throat> του μεταφραστικού έργου. Τα τιμολόγια. Δεν το θεωρώ αυτό χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, που είναι ένα στόχο για εμά παρόλα αυτά. Το ίδιο νιώθω για τη συμφωνία που έχει υπογράψει η ΕΟΚΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λίγους μήνες ε, τώρα για ανταλλαγή ε, κάποιων κτηρίων με το Φαν Δεν κατάλαβα αυτό για το Μοντουάι και το ε, Τρέβ. Χάνουν 10.000 τετραγωνικά μέτρα συν την ανακαίνιση ενός κτηρίου που στη χειρότερη των περιπτώσεων μπορεί και να περιέχει και αμίαντο. Άρα στο μέλλον νομίζω ότι οι συμβουλευτικές επιτροπές θα πρέπει να κάνουν μια εξωτερική μελέτη αντικτύπου και μετά να υπογράψουν ε, την οποιαδήποτε διοργανική συμφωνία. Και για την παρενόχληση, το ανέφερε ο εισηγητής στο θέμα αυτό, για περιπτώσεις ε, παρενόχλησης το 2018 στην ε, ΕΟΚΕ. Νομίζω ότι είχε καταθέσει προσφάτως η Όλαφ την έκθεσή της, όπου όπως λέει ο εισηγητής δεν γνώριζε ότι ίσως υπήρχε αντίγραφο εμπιστευτικό ε, στη διάθεση της Προέδρου. Και συμφωνώ και εγώ ότι αν υπάρχει αυτή η μυστική έκθεση και την έχει πρόεδρος να την πάρουμε και εμείς. Πριν λήξει προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη το περιεχόμενο αυτής της έκθεση και αν δεν μπορεί η πρόεδρο να μας ε, το δώσει η γραμματεία. σε ό,τι αφορά την ιδιωτική χρήση οχημάτων, ε, και αυτό θέλω να το τονίσω, για τις επιτροπές και κάτι άλλο. Θα πρότεινα να τροποποιηθεί η διατύπωση της έκθεσης ε, για τις ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης ό,τι αφορά την, πολιτική, την κτηριακή πολιτική, γιατί δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ολιβιέ Σαστέλ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ με τη σειρά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον Τόμας, ε, για τη δουλειά του. Θεωρώ ότι οι διάφορες εκθέσεις δεν ε, δημιουργούν κάποιο πραγματικό προφανές πρόβλημα σε εμάς τουλάχιστον και το μόνο που θα ήθελα είναι να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποια σημεία. Και πάλι στη διαδικασία απαλλαγής ε, όπως και σε προηγούμενα χρόνια πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ανάγκη να προχωρήσει η ψηφιοποίηση σε όλα τα θεσμικά όργανα. Πρέπει αυτό νομίζω να είναι μια εγκάρσια παρατήρηση για την ψηφιοποίηση δηλαδή και σε σχέση με όλα τα θεσμικά όργανα. Επίσης, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να προτείνουμε γιατί είναι διαφορετικέ οι διαβαθμίσει. να υπάρχει μια πολιτική ανθρώπινου δυναμικού οποία να είναι πιο μακροπρόθεσμη σε ό,τι αφορά το φύλλο, ε, τα άτομα με αναπηρία, ε, τι προοπτικέ εξέλιξη σταδιοδρομία, ε, ισορροπία επαγγελματικού ιδιωτικού βίου. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημείο στο οποίο θα δίναμε οριζόντια έμφαση στο σύνολο των εκθέσεων για τα θεσμικά όργανα. Το ίδιο θα μπορούσα να το είχα πει και το πρωί για άλλες ε, περιπτώσει απαλλαγή. ισχύει για το ότι νομίζω ότι πρέπει να εξακολουθήσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία απαλλαγή. Αν θέλουμε να έχουμε στο έτος νη συνένα τα αποτελέσματα της απαλλαγής και όχι στο τέλος του έτους νη συν δύο. Αυτή είναι μια γενική παρατήρηση. Τώρα, κάποιες ειδικέ παρατηρήσεις ό,τι αφορά το ελεκτικό συνέδριο πρώτα απ' όλα. Να πω ότι σίγουρα πρέπει να κροτήσουμε το έργο του. Κάπου γίνεται λόγο για αύξηση 10% στο στατιστικό δείγμα. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη διαφορά θα κάνει αυτό. Εγώ θα ήθελα να εστιάσει το ελεκτικό συνέδριο στους τομείς που ξεκάθαρα εντοπίζονται γνωστά προβλήματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τη δειγματοληψία. Μιλάμε χάρη για τα ποσοστά σφάλματος σε διάφορους τομείς δραστηριότητα, έρευνα, ανάπτυξη, άγκρη, ρέγγιο. Νομίζω αυτό θα ήταν πιο σκόπιμο. Σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερική πράγματι Μπορώ και εγώ να αναγνωρίσω ότι για την Task Force Stratcom έχουμε αύξηση του προπολογισμού, αλλά θα θέλαμε εν λόγω προπολογισμό να χρησιμοποιηθεί κυρίως για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, αλλά και για τη δημιουργία αυτού του Ινστιτούτου για μελλοντικού διπλωμάτες. Νομίζω ότι και αυτό το Ίδρυμα χρειάζεται χρηματοδότηση. Χαιρετίζω και εγώ την ε, προσπάθεια να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και σύσφυξη σχέσεων μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και ελπίζω όπως και εσείς ε, να έχει αίσιο πέρας να είναι πιο επικοδομητική, θετική η συνεργασία μας σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Έρχομαι στο δικαστήριο. Εδώ θα ήθελα να γίνει έτσι ένας πιο γενικός προβληματισμός σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας ε, των ασκούμενων, των σταζιέρ. Επίσης, η έκθεσή μας θα μπορούσε να είναι πιο συγκεκριμένη και να αναφέρεται ε, στο πρόβλημα της χρήσης ε, των επίσημων, των υπηρεσιακών οχημάτων και των οδηγών από το δικαστήριο, γιατί εκεί βλέπω κάποια πράγματα που πρέπει να τα ε, επισημάνουμε. Και σε ό,τι αφορά τον ε, Ευρωπαίο διαμεσολαβητή, διαμεσολαβήτρα στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει εκεί να καταρτιστεί ένα πραγματικό πρόγραμμα για τη συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου και ένα πιο μακρόπνο πρόγραμμα ε, εργασίας ε, για το θεσμό αυτό. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ολιβιέ. Ο κύριος Έξα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για το σχέδιο έκθεσης, ιδιαίτερα πλήρες και συμφωνώ με τις περισσότερες από τις συστάσεις που κάνετε. Ωστόσο, ως κοιόδης εισηγητής θα ήθελα να προσθέσω κάποια σημαντικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν, πιστεύω, πρώτα απ' όλα. Όσον αφορά το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει εδώ πέρα να αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής, καθότι το Συμβούλιο αποφάσισε να μην συνεργαστεί μαζί μας και μας ανησυχούν ιδιαίτερα οι εικασίες που έχουν γίνει για σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο των, της διαπραγμάτευσης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, σύγκρουση συμφερόντων από συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ πέρα να επιταχυνθούν οι έρευνες που έχουν ξεκινήσει και μάλιστα να ενημερωθεί για τα πορίσματα των ερευνών αυτών και σε κάθε στάδιο της έρευνας του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσον αφορά τώρα την Επιτροπή των Περιφερειών. Θέλουμε να τονίσουμε ότι μετά από 20 χρόνια όπου δεν έχουμε ακόμα επιλύσει την εσωτερική έρευνα που γίνεται όσον αφορά έναν μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Στα τέλη Δεκεμβρίου Προσπαθήσαμε να έχαμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά και πάλι δεν μας δόθηκαν απαραίτητες πληροφορίες. Θεωρούμε ότι αυτές θα πρέπει κάθε φορά να δίνονται στα πλαίσια της διαφάνειας. Η Επίτροπη των Περιφερειών λοιπόν μετά από 20 χρόνια θα πρέπει να αναγνωρίσει το ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή και θα πρέπει να ζητήσει δημόσια ουσιαστικά συγγνώμη για την κακοδιαχείριση και να θεσπίσει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει μελλοντικού μάρτυρε δημοσίου συμφέροντο. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε εμεί να χορηγήσουμε απαλλαγή. Πάντω, όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωση θα πρέπει να εγγυώνται το ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας, δίνοντας σε όλους τους εμπλεκόμενους διακόπτη πρόεδρο. Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρο. πρόεδρος. Τα θεσμικά όργανα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δίνουν στους Ευρωπαίους πολίτες την απαραίτητη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα καθώς επίσης και στις δραστηριότητές τους ακόμα και στις αποστολές που έχουν, στις συναντήσεις που έχουν με ομάδες πιέσεων, λόμπι κτλ. Θέλουμε επίση να τονίσουμε τι προσπάθειε που έχουν καταβάλει τα θεσμικά όργανα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια. Και θα θέλαμε να θαρρύνουμε τα θεσμικά όργανα να χρησιμοποιήσουν ανοιχτέ πλατφόρμε και να εγγυώνται κάθε φορά την προστασία τη ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων πολιτών ένας κοινό τώρα κώδικα διοντολογία. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Κάθε θεσμικά όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωση θα πρέπει να ακολουθεί την ευρωπαϊκή πολιτική κατά της παρενόχλησης, θα πρέπει να έχει ένα πλαίσιο προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντων και θα πρέπει σε κάθε φορά, κάθε φορά να αποφεύγει οποιαδήποτε περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ε, να καταβάλουν όλα τα θεσμικά όργανα συγκεκριμένες προσπάθειες και να έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη μείωση του οικολογικού τους αποτυπώματος και να συμβάλλουν δραστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ που λάβατε υπόψη και τους διερμηνείς. Δεν μπορούν και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους αν μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστούμε. Θα ρωτήσω τώρα αν έχει κάποια άλλη ομάδα σχόλια, VCR, GUE. Ε. Δεν βλέπω να θέλει κάποιο το λόγο. Θα δώσω το λόγο στη Λάρα Βόλτας. Ευχαριστώ πολύ. Να πω δύο λόγια για το Συμβούλιο. Ίσως θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και ένα σημείο που θα αναφέρεται στα προβλήματα του κτίριου Europa. Τώρα το κτίριο έχει ολοκληρωθεί, όμως στο παρελθόν υπήρχαν κάποιες κατηγορίες για εργάτες που δούλευαν χωρίς σύμβαση, χωρίς ασφάλιση. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε και σε άλλες εφημερίδες, πάντως εγώ το διάβασα σε βελγική εφημερίδα πέρυσι. Και η πολιτική μου ομάδα έχει αυτή την ερώτηση λοιπόν. Θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Έπειτα, σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο, έχει να κάνει με τις ε, χορηγίες του. Ε, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω, ε, γιατί διάβασα πρόσφατα πως η Κροατία έχει επίσημο χορηγό ένα βενζινάδικο. Και Μάλιστα διάβασα και ότι Συμβούλιο και Προεδρία δεν έχει καμία διαφορά, το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ πέρα βέβαια κινδυνεύει η φήμη μας. Αν συνεχίσουν να υπάρχουν τέτοιες χορηγίες ε, θα κάνει πολύ κακό στο όνομά μας. Γι' αυτό λοιπόν ε, νομίζω πως η Επιτροπή μας θα μπορούσε να θίξει αυτό το θέμα στην έκθεση της. Ε, νομίζω πως πρέπει να σταματήσουν αυτές οι χορηγίες ή τουλάχιστον να συμπεριλάβουμε το σημείο αυτό σε σύσταση στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο οποίος θα πρέπει να απαντήσει στο Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθο τον Απρίλιο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ωραία. Θα δώσω τώρα ξανά το λόγο στον Τόμα Σεντόφσκι. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί σκιώδεις εισηγητές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά σας Φαίνεται ότι γνωρίζετε σε βάθος το περιεχόμενο της έκθεσης και θα ήθελα να προτείνω να χαρακτηρίσουμε την έκθεση αυτή ως την καλύτερη έκθεση αυτής της χρονιάς. Εξαιρετική δουλειά κάνατε όλοι και νομίζω πως θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο μέλλον. Θα αποτελέσει έμπνευση αυτή η έκθεση. Είμαι ανοιχτό σε όλες ε, τις ε, τροπολογίες σας, να τις συζητήσουμε, να δούμε τι θέλετε να προσθέσω και να πω για το Συμβούλιο ότι στην περίπτωση αυτή θεωρώ πως ο διάλογος είναι ανοιχτός και να ευχαριστήσω τον κύριο Βέλε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το γραφείο της κυρίας Χολμάιερ γιατί έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μας στηρίξατε στις διαπραγματεύσεις και ελπίζω να βρεθεί μια λύση. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους ευρωβουλευτές και για τα κράτη που εκπροσωπούμε. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί μια λύση για αυτήν την ιστορία που πλέον κλείνει δεκαετία. Και κάθε χρόνο ακούμε τα ίδια. Ότι το Συμβούλιο δεν είναι έτοιμο ε, να συμμετάσχει στη διαδικασία απαλλαγή, έχουν ακουστεί επικρίσεις, ότι δεν είναι έτοιμο για διάλογο, όμως νομίζω πως τώρα έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσει επιτέλους αυτός ο διάλογος και να δείξουμε ότι είμαστε πραγματικά έτοιμοι να βρούμε μια λύση. Αυτά από μένα. Καλό υπόλοιπο μέρα. glaube, Νομίζω πως ε, θα παραμείνουμε στην τζίτα σε ό,τι αφορά τη συζήτηση με το Συμβούλιο. Θα δούμε αν θα συμφωνήσουμε. Ελπίζω να συγκλίνουμε περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Ευχαριστώ ξανά όλους εσάς που έπρεπε να ασχοληθείτε και με τα άλλα όργανα τόσα πολλά. Υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια για αυτό το σημείο της σημερισίας διάταξης. Όχι. Να κοιτάξω λίγο και στα δικά μου χαρτιά, να δω σε ποιο σημείο περνάμε. Απαλλαγή 2018. Ε, Νομίζω πως πρέπει να διακόψουμε, διότι δεν έχουν έρθει οι συνάδελφοι για τα επόμενα θέματα, οι συγητές. Δεν έχω τους συγητές για τις κοινέ επιχειρήσεις εδώ. Ήσασταν πολύ γρήγοροι. Ίσως ε, υπάρχει κάποιο σύμβουλος από το ECR για να μας ενημερώσει, να δούμε αν θα έρθουν σύντομα, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να διακόψουμε. Α, Βλέπω ότι η γραμματεία εδώ κάνει κάποιες προσπάθειες. Ξέρετε, χωρίς εισηγητή δεν μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα αυτό. Ωραία, θα διακόψουμε για λίγο μέχρι να έρθουν οι εισηγητές. Τόμας, θέλεις κάτι να πεις? Για 10 λεπτά λοιπόν διακοπή. So, sorry very much. The 10 minutes are over. Λοιπόν, πέρασαν τα 10 λεπτά και πρέπει να συνεχίσουμε με το θέμα για τις κοινέ επιχειρήσεις. Ζητώ συγγνώμη από τους ε, εισηγητές που βιαστήκαμε τόσο πολύ και έπρεπε να σας φωνάξουμε να έρθετε πριν την ώρα σας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μπροζίνσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Προφανώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, γιατί όταν επεξεργαζόμουν τις εκθέσεις αυτές, έλαβα πραγματικά πολύτιμη βοήθεια από εσά και από τη γραμματεία της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια και τους συμβούλους μας, την Καμίλα Συντίσκα που κάθεται στα αριστερά μου, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. «14 Νοεμβρίου του 2018 το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο δημοσίευσε μία κοινή ενία έκθεση όσον αφορά τις κοινέ επιχειρήσεις. και εκεί επιβεβαιώθηκε η αξιοπιστία και η κανονικότητα των λογαριασμών όλων των κοινών αυτών επιχειρήσεων. Η έκθεση αυτή η ενία επίσης επιβεβαιώνει την αξιοπιστία, την νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των οικονομικών συναλλαγών και αναφέρεται στην έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου ότι υπήρξε μια καθυστέρηση όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος Horizon 2020. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο στην εκθεσή του αναφέρει ότι η εφαρμογή του προηγούμενου προγράμματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αναφέρεται επίσης στο σημείο 4η μία σχετική μνήμα στις καθυστερήσεις αυτές. Τώρα στις α, εκθέσεις του 2018 αναφέρονται και οι κοινέ επιχειρήσεις και προφανώς σήμερα θα πρέπει να συζητήσουμε για το αν μπορούμε να χορηγήσουμε απαλλαγή σε σχέση πάντα με το οικονομικό έτος 2018, σε σχέση με τον προπολογισμό των κοινών αυτών επιχειρήσεων, σε σχέση με την στρατηγική προσλήψεων, σε σχέση με τη στρατηγική δημοσίων προμηθειών, σε σχέση με τη στελέχωσή τους και ούτω καθεξής και σε σχέση με τις υποχρώσεις που έχουν υποβολή εκθέσεων και εσωτερικού ελέγχου πάντα για το έτος 2018 βέβαια. Τα προηγούμενα οικονομικά έτη δεν ετέθη να αμφιβόλο καθόλου η διαδικασία απαλλαγή. Μόνο το 2014 είχαμε συναντήσει κάποια προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι η θετική αυτή τάση που είχαμε και τα προηγούμενα έτη θα συνεχιστεί και φέτος. Εν γέννη πάντως, η κατάσταση σε σχέση με τις κοινέ επιχειρήσεις τελεί από ένα θετικό καθεστώς παρακολούθησης και δεν υπάρχει κανένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν επιμέρους μονοπτυχές, τις οποίες θα ε, πρέπει να προσέξουμε λίγο περισσότερο ως εισηγητές και επί των οποίων θεωρούμε ότι υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον κύριο Λεγκούτκο να αναφερθεί ε, πιο επισταμένος στις πτυχές εκείνες όπου θεωρούμε ότι υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης. Ο κύριος Λεγκούτκου λοιπόν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όντως θα ήθελα να θίξω μερικά σημεία. Πρώτον, όσον αφορά το IMI 2. Το 2018 το ποσοστό στελέχος ήταν υψηλό, 20%, ιδιαίτερα υψηλό λοιπόν, και είχαμε φτάσει σε ένα συνολικό ποσοστό 60% και αυτό διότι είχαμε τέσσερις νέες περιπτώσεις αδειών ασθένεια σε σύνολο 8, τέσσερις νέες περιπτώσεις για το 2018. Και βλέπουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο για το έτος 2018 και για την κοινή αυτή επιχείρηση είχαμε προβλήματα όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους της κοινής αυτής επιχείρησης, που ενδεχομένω να μην καλύπτονταν. Είδαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωση αυτή συμβασιούχοι προσωρινά απασχολούμενοι 9,6% του συνόλου προσωπικού για το 2018 πάντα. Αυτά όσον αφορά το IMI 2. Τώρα, όσον αφορά τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοπορία, για την κοινή αυτή επιχείρηση εντοπίσαμε, μάλλον το λεπτικό συνέδριο, εντόπισε δυναμίες όσον αφορά τις δημόσιε δημόσιες προμήθειες για διοικητικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και οι εισφορές σε μετρητά που ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο ευρώ και για τα οποία δεν υπήρχε συγκεκριμένο τιμολόγιο προτού α, θεσπιστεί το έξω. Τώρα όσον αφορά το Clean Sky 2. Σε σχέση με το οικονομικό έτος 2017, το 2018 αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα ποσοστά προσωπικού ήταν ε, υψηλά για τους συμβασιούχους και τους προσωρινά απασχολούμενους και είδαμε ότι για το προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό είχαμε μια αύξηση της τάξης του 17% και ε, για τους συμβασίουχους διπλασιάστηκε το προηγούμενο ποσοστό. Όσον αφορά τώρα την κοινή επιχείρηση βιομηχανικών βιοπροϊόντων, από τα 182.500.000 εισφορές σε μετρητά που θα γινόντουσαν από τις βιομηχανίες των κρατών μελών προς την κοινή αυτή επιχείρηση για την κάλυψη του κόστους μόνο 800.000 ευρώ είχαν καταβληθεί μέχρι τα τέλη του 2018 και επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στα τέλη του 2018 να μειώσει τον προπολογισμό του 2020 για την κοινή αυτή επιχείρηση κατά 205 εκατομμύρια ευρώ, από 205 εκατομμύρια ευρώ σε 140. Με συγχωρείτε, μπέρδεψα λίγο τα μηδενικά, λέει ο, ο ...205 εκατομμύρια και φτάσαμε στα 140 εκατομμύρια. Αυτή ήταν η μείωση από 205 στα 140 εκατομμύρια. Και ενδεχομένω να μην καταφέρουμε εδώ πέρα να έχουμε την απαιτούμενη συνεισφορά από τι βιομηχανίε μέχρι το τέλο τη εντολή αυτή τη κοινή επιχείρηση. Τώρα, όσον αφορά την κοινή επιχείρηση ITER, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας Σύνδεξης. Η κοινή αυτή επιχείρηση αποτελεί ουσιαστικά ένα διεθνές ε, πρόγραμμα και ουσιαστικά παρουσιάζει τις περισσότερες προκλήσεις, τις οποίες ε, έχουμε προσπαθήσει να περιγράψουμε. Προσπαθήσαμε εδώ πέρα να επανυπολογίσουμε το κόστος το οποίο απαιτείται όσον αφορά την φάση οικοδόμησης 12 δισεκατομμύρια ευρώ από 6 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια που ήταν ο αρχικός προβλεπόμενος προπολογισμό. Πραγματικά μπορώ να πω ότι μου προκαλούν ήλιγκ όλα αυτά τα μηδενικά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Εγκρίθηκε αυτό ο αρχικό προπολογισμό από το Συμβούλιο του 2018 και δεν περιλαμβάνει το προπολογισμό έκτακτη ανάγκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει ότι θα μπορούσαμε να είχαμε μία περίοδο έκτακτη ανάγκη έω 24 μήνε, ακριβώ επειδή υπήρχαν καθυστερήσει στην εκτέλεση του προγράμματο αυτού. Τώρα, τον Νοέμβριο του 2016, το Συμβούλιο της Κοινής Επιχείρησης ΣΥΤΕΡ ενέκρινε μία νέα γραμμή βάσης που αξιολογεί τα επιτεύγματα από το πρώτο πρόγραμμα πλάσματος και αρχίζει την διαδικασία κατασκευής του 2025 με προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία το 2035, ενώ η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν το 2020. Το 2018 υπήρχαν κάποιες αδυναμίες όσον αφορά την κατάρτιση του προπολογισμού και απαιτήθηκαν περισσότερες πιστώσεις πληρωμών για το 2017 και το 2018 που υπερέβησαν τις αρχικές, αρχικά προβλεπόμενες πιστώσεις πληρωμών. Προέκυψαν επίσης και κάποια άλλα εσωτερικά ζητήματα. Τον Ιανουάριο 2018 το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό, μάλλον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ασχολήθηκε με το σύστημα προσλήψεων το οποίο είχε εγκρίνει η κοινή αυτή επιχείρηση. Και το δικαστήριο ε, ε, εντόπισε τελικά, ακύρωσε τη διαδικασία την οποία είχε αρχικά εγκρίνει η κοινή αυτή επιχείρηση όσον αφορά το σύστημα προσλήψεων. Και νομίζω ότι θα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη ιδίω για τις δραστηριότητες εκείνες οι οποίες θα αναλυφθούν από το 2020 και μετά. Με την άδειά σας τώρα, κυρία Πρόεδρε, και ο κύριο Μπριζίνσκι θα ήθελα να σας δώσει κάποιες περαιτέρω πληροφορίες. Να ξαναπάρει ο κύριο Μπριζίνσκι τότε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη κοινή επιχείρηση, Shift to Rail. Το 2018 ένα από τα μέλη της κοινή αυτής επιχείρησης έγινε ουσιαστικά θηγατρική επιχείρηση που βρίσκεται υπό το καθεστώς ιδιοκτησίας της ιδρυτικής εταιρείας. Και αναφέρομαι εδώ πέρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις που έλαβε η κοινή αυτή επιχείρηση. Όσον αφορά τώρα τις κοινέ επιχειρήσεις, ξέρετε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο επί ε, στα πλαίσια του οποίου δεν προβλέπονται συγκεκριμένε λύσεις όταν μια συγκεκριμένη επιχείρηση ουσιαστικά εξαγοράζεται από ένα από τα μέλη του βιομηχανικού αυτού κονσόρσιουμ. Πώς μπορούμε με άλλα λόγια να διασφαλίσουμε ότι όντως θα υπάρχει μια ισότιμη εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση της κοινή επιχείρησης Caesar είχαμε μια ειδική έκθεση από το λεκτικό συνέδριο όσον αφορά την επίτευξη λύσεων στην περίπτωση αυτή. Φαίνεται ότι τα περισσότερα προγράμματα τότε θα πρέπει να χρηματοδοτούνται χωρίς να υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπήρχαν συγκεκριμένες αδυναμίες. Παρ' όλα αυτά δεν εντοπίστηκαν Επιπτώσει όσον αφορά τη διαχείριση της ενέργεια κυκλοφορία, όσον αφορά έπειτα τις κυψέλε καυσίμου και το υδρογόνο. Στην κοινή αυτή επιχείρηση δεν έχουμε να κάνουμε συγκεκριμένε παρατηρήσει ενδεχομένω για τον προπολογισμό του 2018 και το πώ αυτό συνδέεται με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Εδώ πέρα είχαμε κάποιε καθυστερήσει όσον αφορά τι αποζημιώσει για συγκεκριμένα προγράμματα που ήταν σε εξέλιξη και είχαμε περίπου 79,6% υπέρβαση προπολογισμού όσον αφορά συγκεκριμένα προγράμματα. Θεωρούμε παρόλα αυτά ότι θα πρέπει να μπορούμε για όλες αυτές τις κοινέ επιχειρήσεις να χορηγήσουμε απαλλαγή. Σας ευχαριστούμε και είμαστε θέσεις για τυχόν ερωτήσεις στα πλαίσια της συζήτησης. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την καταπληκτική σας δουλειά. Να δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Αγαπητέ Πίπερ, από πλευρά ΣΕΛΚ, είστε ο πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συζητητές. Εμείς ε, συμφωνούμε και θα χορηγήσουμε τις απαλλαγές αυτές, αλλά έχουμε τρεις παρατηρήσεις. Θα καταθέσουμε τροπολογίες για τα εξής. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τις κοινέ επιχειρήσεις, κάνουν πολλά θετικά, δημιουργούν προσθέμενη αξία στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι τόσο προβεβλημένες. Αν είμαι στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, μόνο ξέρω τι κάνουν αυτές οι κοινέ επιχειρήσεις. Και είναι κρίμα για τα χρήματα των φορολογουμένων. Επομένως θα πρέπει να έχουμε επικοινωνία, να επικοινωνήσουμε προς τα έξω για τα αποτελέσματα των κοινών αυτών επιχειρήσεων. Όταν ε, ερευνούμε κάποια θέματα, όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε συνέργειες και να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και αν τελικά τα πετυχαίνουμε όλα αυτά, πρέπει και η κοινή γνώμη να ενημερώνεται. Και αυτό ισχύει ε, για όλες αυτές τις κοινέ επιχειρήσεις. Και πραγματικά σε ό,τι αφορά ε, το πόσο γνωστά είναι τα αποτελέσματα του έργου αυτών των επιχειρήσεων, πρέπει να πω ότι είμαι απογοητευμένο. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, είναι μια τεχνική παρατήρηση. Νομίζω ότι θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες. για κάποια θέματα και σε ό,τι αφορά την ε, διατύπωση ε, θα καταθέσουμε επίσης ε, τροπολογίες για κάποια ζητήματα που αναφέρονται έτσι με πολύ αρνητικό τρόπο και θα θέλαμε να δώσουμε έτσι μια πιο θετική απόχρωση. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ. Λάρα Βόλτες, στη θέση της κυρίας Γκραπίνη. Ευχαριστώ. Πράγματι, κυρία Γκραπίνη, είναι σκιώδης. Μου έδωσε μια σημείωση εδώ να διαβάσω, ένα σημείωμα. Αλλά επειδή είναι τρεις σελίδες, δεν θα τα πω όλα. Σίγουρα ήθελε να είναι πάρα πολύ ε, αναλυτική, αλλά δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα, δεδομένου του χρόνου. Θέλει λοιπόν να αναφέρει ότι τα αποτελέσματα των κοινών επιχειρήσεων το 2018 ήταν θετικά και μπόρεσαν να ξεπεράσουν κοινέ επιχειρήσει τις προκλήσεις. Θέλω να ευχαριστήσει τους κοιότες για τις ε, εκθέσει τους, θα συνεργαστεί μαζί τους και λέω τα αποτελέσματα των ελέγχων για τις κοινές επιχειρήσεις από πλευράς ελεγκτικού και η ε, εκθέσεις δείχνουν ότι υπήρξε νομιμότητα και κανονικότητα. Θετικά όλα αυτά εκτιμώνται για το 2018. Ε, συνιστά βελτίωση κατάσταση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Έπειτα κύριε Γκραπίν κάνει κάποια σχόλια για ορισμένα από τις κοινέ αυτές επιχειρήσεις. Κάποια έχουν ήδη αναφερθεί, άρα δεν θα τα αναφέρω. Για το shift του rail, λέει ότι ναι, μεν υπήρξε πρόοδο για την επίτευξη των στόχων από την κοινή αυτή επιχείρηση, αλλά ή και δεν έχω καταλάβει ακριβώ, πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόσει τη στρατηγική για την καταπολέμηση απάτη ε, μέχρι το 2020. Δεν εστάλει κάποιος φάκελο στην Όλαφ για έρευνα μετά από τις ε, έρευνε που έγιναν και σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, δεν γίνεται... Ε, δεν είναι επαρκή τα όσα προβλέπονται στο πλαίσιο των διαγωνισμών. Πρέπει να υπάρχει ένα μητρό ενωπημένου κινδύνου και υπήρχαν και τρεις περιπτώσεις ε, ε, για ενδεχόμενη απάτη. Κάποιοι δικαιούχοι πήραν ε, από την εταιρεία κάποια χρήματα και θα πρέπει να αποφευθεί στο μέλλον κάτι αντίστοιχο για καινοτόμα φάρμακα. Υπήρξε ανακύκλωση, αλλά στο προσωπικό ιδίως για τους συμβασιούχους. Και η κατάσταση επιδεινώθηκε γιατί το 18 ήταν 8 ε, άτομα σε μακροχρόνια ερωτική, δηλαδή το μισό προσωπικό λειτουργούσε. Δεν ξέρω αν το έχει ξαναπεί κάποιο αυτό. Για τα βιοπροϊόντα. Δεν είναι θέμα η, η έλλειψη κοινών, ε, μάλλον βασικών δικτών επιδόσεων, αλλά υπάρχει κίνδυνος. Ότι μπορεί κάποιοι στόχοι να μην έχουν ε, ολοκληρωθεί μέχρι την ε, λήξη ισχύω της κοινή επιχείρηση τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, Excel, βρήκε αδυναμίες στη διαχείριση των δημόσιων προμηθειών το ελεκτικό συνέδριο και επίσης ένα άλλο πρόβλημα είναι οι συμβολές της μετρητής. Για το ίτερ υπήρχαν προβλήματα στη διαδικασία σχεδιασμού, του προπολογισμού και λέει ότι για τις πιστώσεις πληρωμών το 2017 και 2018 υπερεύησαν σημαντικά τον αρχικό προϋπολογισμό. Η εταιρεία βέβαια έχει σημειώσει πρόοδο για να πετύχει τους στόχους. Και το σύστημα των προβλέψεων έχει αναθεωρηθεί και θα χρησιμοποιηθεί για το 19 και αυτό είναι θετικό. Θα συνεργαστεί με όλους τους συναδέλφους και θα περιμένει και τις τροπολογίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία σύνοψη. Περνάω τώρα στην Μαρτίνα, η συγγύτρια από την ομάδα Renew. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι του Ελεκτικού Συνεδρίου και των Κοινών Επιχειρήσεων, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ε, συνέχεια που χαρακτηρίζει την έκθεση. Ε, ήμουν εισηγήτρια στην περσινή έκθεση και προς στιγμή νόμιζα ότι διάβαζα την περσινή έκθεση, τη δική μου. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που υπάρχει αυτή η συνέχεια. Θεωρώ πως οι κοινέ επιχειρήσεις το χρειάζονται αυτό. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τις κοινέ επιχειρήσεις για την προστιθέμενη αξία που δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την επιτυχία που έχουν δείξει και την ενότητα που τους χαρακτηρίζει. Είστε πραγματικά εμβληματικές επιχειρήσεις για την Ευρώπη. Χρειάζεται όμως να βελτιωθεί αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος. Ε, δεν φτάνει μόνο να βελτιωθεί η διαδικασία δημόσιων προμηθειών και προσλήψεων, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Όπως αναφέρει και η έκθεση, το ε, ποσοστό σφάλματος που είναι κάτω από το όριο, όμως ε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκε πως η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν ήταν αναγκαία. Οι κοινέ επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να κινητοποιήσουν πρόσθετους πόρους, να δημιουργήσουν συνέργειες και εντός και εκτός ενιαίας αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών. Ορισμένες κοινέ επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν τις πιστώσεις πληρωμών ε, στο πρόγραμμα πλαίσιο 7 θα καταθέσω τροπολογίες που θα έχουν να κάνουν περισσότερο με τις επιδόσεις. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ πολύ ε, για τη δουλειά που κάνατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πέξα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μιλώ εκ μέρους του συναδέλφου που δυστυχώς απουσιάζει. και εκείνη θα καταθέσει τροπολογίες, αλλά δεν θα είναι τίποτα το ιδιαίτερο και το ανησυχητικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Από το ID και την ΚΟΕ e δεν έχουμε νομίζω κάποιον παρόντα που θέλει το λόγο, οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια σε περίπτωση που θέλει να κάνει κάποια καταληκτικά σχόλια στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, έγιναν λοιπόν κάποια τεχνικά σχόλια, να κάνω και εγώ κάποια γλωσσι... κάποιες γλωσσικές παρατηρήσεις. Ε, υπάρχουν τα έγγραφα διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα της Επιτροπής. Υπάρχει και η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου εκεί, καθώς και η τελική έκθεση. Καταληκτικές ημερομηνίε λοιπόν για τροπολογίες. 29 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ψηφίζουμε στην Επιτροπή στις 19-20 Φεβρουαρίου και ίσως στην Ολομέλεια ψηφίσουμε ε, το Μάρτιο, στη δεύτερη Ολομέλεια του Μαρτίου. Περιμένουμε λοιπόν τις τροπολογίες σας και μόλις εκείνες φτάσουν θα διοργανώσουμε ε, συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε ξανά και τους δύο συγητές και ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία με τους σκιώδεις συγητές. Να σας ενημερώσω και για το χρονοδιάγραμμα με τη σειρά μου. Έχετε τις ημερομηνίες στο, στα εγγραφά σας για τις τροπολογίες και όπως είπε και ο κύριος Μπροσίνσκι, για την ψηφοφορία στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Επόμενη συνεδρίαση στις 28 Ιανουαρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6.30 το απόγευμα 29 Φεβρουαρίου 20 Φεβρουαρίου μετά και στις 27 Ιανουαρίου θα γίνει μια τεχνική συνάντηση ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου θα έχουμε διάφορους εκπροσώπους παρόντες και θα μπορείτε να τους κάνετε ερωτήσεις. Σε αυτό το σημείο λοιπόν μπορώ να ολοκληρώσω τη συνεδρίαση και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ich frage einfach 4 um er um äh, ε, ε, θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση των ε, συντονιστών ή δυνατών. Ο Κλαουδίο να ρωτήσει παρακαλώ αν αυτό είναι δυνατό, αντί των 4.30 που προβλεπόταν. Να με ενημερώσετε παρακαλώ. Οπότε παρακαλώ να μείνετε όσοι είστε για τη συνεδρίαση των συντονιστών. Θα χαιρετήσω όλους τους υπόλοιπους και τους συντονιστές θα σας δω οι 4-4.30 το αργότερο. Damit